αυτό η ψηφορία θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο σήμερα σήμερα στη διάλεξη. Έκθεση του συναδέλφου Σμιτ για την ετήσια έκθεση για την φορολογία. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή για 4 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί Επίτροπε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανέλαβα τα καθήκοντα του εισηγητή για αυτή την έκθεση. Πρόκειται για την πρώτη ετήσια φορολογική έκθεση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ του και όλους εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία για αυτό το ενδιαφέρον αλλά δύσκολο θέμα. Προσπάθησα να συμπεριλάβω σχόλια από όλε τι πολιτικέ ομάδε στην έκθεση και νομίζω ότι τελικά καταλήξαμε σε κάποια συνεννόηση. Ελπίζω να τύχει ευρεία υποστήριξη η έκθεση. Η φορολογική πολιτική είναι ένα θέμα που αγγίζει άμεσα τους πολίτες ε, διότι ε, δημιουργεί θετικά και αρνητικά αισθήματα για πολλούς. Υπάρχουν περισσότερες διενέξεις στα πλαίσια της φορολογικής πολιτικής σε σχέση με άλλους τομείς. Πάντοτε αναζητούμε την σωστή ισορροπία. Δεν είναι ε, εύκολο. Πάντως ε, θεωρεί το ε, ως εθνική πολιτική φορολογική πολιτική στο παρελθόν. Όμως ε, έχει παρέλθει αυτός ο χρόνος πλέον. Τα φορολογικά ζητήματα θα πρέπει να παγκοσμιοποιηθούν και να συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της έκθεσης είναι να ερευνήσουμε περαιτέρω τα φορολογικά ζητήματα και να τίνουμε σιγά σιγά προς ενός είδους φορολογική εναρμόνιση. Νομίζω ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η έκθεση επίση. Χρειάζεται μια ενοποίηση κρίση των φορολογικών διατάξεων, ε, διότι η δημοσιονομική κρίση εν μέρει είναι και φορολογική ε, κρίση. Δεν υπάρχει επαρκή συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών και των φορολογικών πολιτικών και αυτό οδηγεί σε βαθύτερη ακόμη κρίση. Επίσης, ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε, όπω αναφέρω μέσα στην έκθεση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα για να προστατεύσει τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και να δημιουργήσει μια ανταγωνιστικότερη Ευρώπη. Δυστυχώ υπάρχουν πολλέ εταιρείε ακόμη ε, και οι πολίτε που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω των φορολογικών κολλημάτων. Πρέπει να άρουμε λοιπόν αυτά τα κολλήματα για να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και να αναπτυχθεί το επιχειρηματικό πνεύμα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μειώσουμε τι ε, φορολογικέ ε, εισφορέ και να βελτιώσουμε με έτσι την κατάσταση στην αγορά εργασία. Ελπίζω μέσα από αυτή την έκθεση να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη για να εγκριθούν οι φορολογικέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και η εισαγωγή του CCTB, του περίφημου δηλαδή τη ενιαία φορολογική βάση για τι εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, ε, κάποιοι που ζουν σε μια χώρα και εργάζονται σε κάποια άλλη υποφέρουν από τη διπλή φορολόγηση. Οι φορολογικέ συμφωνίε για την αποφυγή τη διπλή φορολογία δεν επαρκούν για να αποφευθεί αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν επαρκώς διεξοδικές διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Στην Επιτροπή Αναφορών είχαμε έναν Ιταλό οδηγό φορτηγού που δούλευε και στη Γερμανία και ε, στο ύψος του 60% των εισοδημάτων και από τις δύο χώρες, ενώ θα έπρεπε ε, να πληρώνει μόνο στη Γερμανία 25% και όχι 60%. Βλέπετε τις φορολογικές διαφορές λοιπόν ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ιταλία και παρότι οι φορολογικές ε, αρχές έχουν διαπιστώσει ότι είναι λάθος να συμβαίνει αυτό, δεν έχουν επανορθώσει την κατάσταση ακόμη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε η κοινοτική νομοθεσία, ούτω ώστε να κάνουμε τη διαφορά. Καλωσορίζω λοιπόν την πρόσφατη έγκριση τη ανακοίνωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διπλή φορολόγηση όπου προτείνονται συγκεκριμένα ειδικά μέτρα. Τώρα φοροδιαφύγη, ε, ε, ε, αυτό οδηγεί σε απώλεια εισοδημάτων του ύψου δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να κλείσουμε όλα αυτά τα παραθυράκια που υπάρχουν στην κείμενη νομοθεσία, τόσο ώστε οι πολυεθνικέ εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορούν πλέον να φοροδιαφεύγουν. Οι φιλοδοξίε μα ε, πρόεδρε, αγαπητοί Επίτροποι, θα πρέπει να είναι να ε, υπάρχει σωστά, σωστή ενημέρωση και ένα ε, κρατεό πλαίσιο, τόσο ώστε στο μέλλον να μην πλήττονται ούτε οι πολίτε ούτε και τα εισοδήματα φορολογικών αρχών. Η παράγραφο 11 έχει δημιουργήσει, να πω κλείνοντα, ότι έχει δημιουργήσει μία μικρή σύγχυση και θα αντικαταστήσουμε το κείμενο από την πρόταση του Μπομπάσκη και Καταλίνε από συναδέλφου. Παραθέτω Πιστεύει ότι η ομοσπονδιακή προσέγγιση στα φορολογικά θέματα είναι η βέλτιστη λύση, ούτω ώστε ε, να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για φορολογική διαχείριση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και ε, να επιτύχουμε μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα. Αυτά θα αντικαταστήσουν διατύπωση του άρθρου τη παραγράφου μάλλον 11. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφε κύριε Κοιτάξτε, ε, ήταν σημαντικό αυτό που θέλατε να προσθέσετε, είπατε. Α, σήμερα έχουν χρόνο, αλλά κανονικά δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα λεπτό στο χρόνο αγόρευσή σα. Κασουζάη, πίλτ Πίλ πρώτο. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κατεβάσει αυτή την, ε, προτείνει αυτή την έκθεση όσον αφορά τις ε, φορολογικές πολιτικές και νομίζω ότι και αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Αλλά έτσι θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε εκατομμύρια ευρώ τα οποία τώρα χάνονται. Πάρα πολλές χώρες δεν έχουν μπορέσει να συμμετάσχουν πλήρως στην ενιαία αγορά. Αυτή τη στιγμή είναι εθνική αρμοδιότητα η φορολογική πολιτική. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη διαφάνεια, αλλά και συγκρισιμότητα στις ε, ε, πολιτικές αυτές. Και κυρίως επιτονίζω την συγκρισιμότητα των φορολογικών πολιτικών των μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταπολεμήσει την ε, φοροδιαφυγή, την απάτη, αλλά να αποφευθεί διπλή φορολόγηση. Πέραν του όσα, να κινητοποιηθούμε όλοι. Ευχαριστώ, συνάδελφε ε, Γκάλπελτ. Ο συνάδελφο Ελκαραντού έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Σμίτε για την εξαιρετική αυτή έκθεση και τη συνεργασία που είχαμε. Η κρίση χρέους που ζούμε στην Ευρώπη μας υποχρεώνει να ε, επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουμε την οικονομική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φορολογικά ζητήματα. Θα πρέπει να αναμφισβήτητα να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και γενικότερα σε επίπεδο Ένωση. Ε, η ομάδα μου πιστεύει ότι αυτό συνεπάγεται δικαιότερη φορολόγηση, αποφυγή της φοροδιαφυγής στο ιστορικό της Ένωσης, αλλά και εκπόνηση μιας κοινωνική στρατηγικής ε, ως προς τα, τρίτα κράτη-μέλη. Ε, γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να συναυθούν ε, ταχύτατα διμερείς συμφωνίες όπως με την Ελβετία. Αλλά αυτό που προκρίνουμε είναι μια σφαιρική γενικότερη προσέγγιση, δηλαδή συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία. Ο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την εναρμόνιση τη φορολογική βάση ε, για τι εταιρείε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, κύριε Αλκαρατούη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο βασικός σκοπός κάθε φορολογικού στήματος λέει ο αγορητής μιλάει εντύπωση για την Παραντίκα. Συγγνώμη με δικαπτή πρόεδρος. Η κυρία Βιλπά Παραντίκα έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι διότι υποστηρίχθηκε αυτή η έκθεση από το Κοινοβούλιο και πάμε τώρα για έναν φεντεραλισμό, μια ομοσπονδιακή ούτως η λύση για τις φορολογικές πολιτικές γιατί το, το, όπως υπάρχει κοινή πολιτική για τις δαπάνες θα πρέπει να υπάρχει για τα έσοδα έτσι να ξεπεράσουμε το, το πρόβλημα του ελλείμματος και να πάμε σε πιο παραγωγική οικονομία επίσης είναι πάρα πολύ ε, βασικό το, το να δούμε τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να στηριχθούν οι περιφέρειες που έχουν φορολογικές αρμοδιότητες και να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες σε αυτούς που τις ζητούν και σύμφωνα με τις αρχές ε, της ε, χρηματοοικονομικής σταθερότητας υπάρχει σχετική δέσμη μέτρων και θέλουμε να υπάρχει εναρμόνιση αλλά θέλουμε να υπάρχει ισότητα μεταξύ περιφερειακών και κρατικών φορολογικών πολιτικών διότι αυτή τη στιγμή Αυτά τα μέτρα τα φορολογικά που επιβάλλονται σε κάποια κράτη-μέλη ε, ε, ε, επικρίνεται η βασική κυβέρνηση γιατί εφαρμόζει τα ίδια μέτρα στην περιφερειά της. Συμφωνώ με τον κύριο Σμιτ ότι η φοροδιαφυγή ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι κάτι πρέπει να γίνει ε, για τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών φορολογικών πολιτικών. Δεν πιστεύω ότι η εναρμόνιση είναι η καλύτερη ρότα. Τα κράτη-μέλη ε, δεν το επιθυμούν εξάλλου. Αντίθετα, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ε, επεξεργαστούμε ε, κοινά λογιστικά ε, συστήματα και πρότυπα, υποδείγματα τιμολογίων που θα γίνονται δεκτά ως παραστατικά από διάφορες φορολογικές αρχές σε όλα, στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Πέραν τούτου θα μπορούσαμε επίσης να συμφωνήσουμε επί μιας ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείε. Πιστεύω πώς ε, θα παραμείνει εθνική αρμοδιότητα η φορολογική πολιτική για πολύ καιρό. Ευχαριστώ, συνάδελφος Λούχαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα... Ήθελα να σας πω ότι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 500 εκατομμυρίων πολιτών ο καθένας θα πρέπει να ωφελείται από τα δικαιώματα του βάση του κοινοτικού δικαίου. Δυστυχώς οι διακρατικές δραστηριότητες είναι πάντα δυνατές. Αυτό είναι άδικο και υποσκάπτει τις αρχές της ενιαίας αγοράς. Για να αυξηθεί η κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε νομίζω ειδικού κανόνες για τους διαμεθοριακούς ε, εργαζόμενους ε, που θα λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για την ε, σχέση μεταξύ των ε, φορολογικών ε, συστημάτων και συστημάτων κοινωνική ασφαλής των κρατών μελών γιατί θα πρέπει να έχουμε μια εναρμόνιση των εθνικών προτύπων που είναι απαραίτητη για τις εταιρείε και τους πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τη σήμερα ημέρα η χρηματοοικονομική κρίση μας έχει οδηγήσει σε αύξηση του κρατικού ή δημοσίου χρέους. Επομένως, η κοινωνική πολιτική τώρα είναι πιο σημαντική παρά ποτέ. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να καλύψουμε τις προσδοκίες των Ευρωπαίων, για να χρειάζεται κάποιο είδους παγίωση ε, τις φορολογικές πολιτικές. Αλλά θα πρέπει όμως βέβαια η φορολογική βάση να είναι δίκαιη. Να είναι προοδευτικά τα κλιμάκια σε σχέση με το ποιοι πληρώνουν και έτσι θα διηγηθούμε πιο εύκολα στην οικονομική ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε εις μέτρα που θα σταματήσουν την φοροδιαφυγή. Άρα χρειάζεται η διαφάνεια. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ο συνάδελφος Φεγιό έχει το λόγο. E, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον εισηγητή που, που αυτό το έργο, διότι τώρα πρόκειται εδώ για ένα θέμα άκρο ιδεολογικό. Έχουμε διάφορε αναλεκτικές. Ο κύριος Όλε Σμιτ μπόρεσε έτσι να οδηγήσει σε, κάποια συνένεση που σημειώθηκε. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την φορολογική εναρμόνιση και για την φορολόγηση των εταιριών, για την φορολογική βάση που επιλέγουν τα κράτη-μέλη και εφαρμόζουν προς το παρόν, μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Ω προ τον φορολογικό ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τι τρίτε ε, χώρες. Ε, έχει καθοριστική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ανταγωνιστικά φορολογικά συστήματα έτσι ώστε να επισύνουν πλούτο επενδύσεις ε, που τόσο χρειαζόμαστε λόγω της κρίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Κρέτικα, όχι. Funcția principală a sistemelor fiscale este de a finanța servicii. Πρόεδρε, η φορολογία χρηματοδοτεί μεταφορές, παιδεία, ε, ε, γενικά τις κρατικές υπηρεσίες και επίσης ε, βοηθάει στην κατανομή του πλούτου. Οπότε έτσι θα πρέπει να οδηγηθεί η φορολογία να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, ανταγωνιστικότητα και να βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε θα πρέπει να μπορούν οι φορολογικέ αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να καλύπτουν τις προσδοκίε των πολιτών και άρα θα πρέπει να συγχυστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και έτσι να αντιμετωπίζεται η απάτη, η φοροαποφυγή, να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και να ισχύει ένα κράτος δικαίου Οπότε θα πρέπει και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα να εντοπίζονται δίκαια Επίση, η ε, ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και καθαριστικών είναι η απάντηση και θα πρέπει να υπάρχει ισότη μεταχείριση. Ευχαριστώ κύριε Τσικάου. Τελευταία η κυρία Μεσέσκου στη διαδικασία Κατσουδιάη. Κύριε Πρόεδρε, η έλλειψη προλογικής πολιτικής πανευρωπαϊκής είναι φραγμός στο να έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Οδηγείται έτσι η κατάσταση σε περισσότερη απάτη και φοροδιαφυγή. Άρα θα πρέπει να αρθούν οι σχετικοί φραγμοί και να έχουμε έτσι περισσότερη διασυνοριακή δραστηριότητα. Πάρα πολύ σωστό είναι το ότι έχει συγκροτήσει η ομάδα εργασίας για να έχουμε αποφυγή διπλής φορολογίας. Έτσι, αυξάνεται το φορολογικό βάρος, πλήσεται η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιες συμφωνίες σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας και έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Έχουμε άλλωστε κάποια πρόσφατα στοιχεία που μας δείχνουν ότι οι επενδύσει έτσι δύναται να αυξηθούν κατά 50% εάν προχωρήσουμε σε τέτοιες συμφωνίε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πεσέσκο. Ολοκληρώνεται η διαδικασία Κασδιάη εδώ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος θα δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπη, κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέτει το θέμα της φορολογικής φορητικής ε, πολύ ψηλά στην μεσαιοδιάταξη όπως φαίνεται και από το σημείο αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σμιτ γιατί η θέτει πραγματικά πολύ ψηλά τον πύχη για εκείνο που θα ακολουθήσουν. νόμο της Κομισιόν, θα ήθελα να χαιρετήσω την ευρεία υποστήριξη των πρωτοβουλίων τη Επιτροπή και οι πολύ αξιόλογες προτάσεις που υποβλήθηκαν για τη μελλοντική μας εργασία είναι επίσης καλόδεκτες. Θα ήθελα να μπω κάπως περισσότερες λεπτομέρειες. Πρώτον, στο σημερινό οικονομικό κλίμα η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφέστατα χρειάζεται μια πιο ε, δραστήρια ε, πολιτική όσον αφορά τον, τόμο, τον ε, τομέα των φορολογικών. Στους στόχους του 2012 η Κομισιόν ε, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό για τα κράτη-μέλη. Βρέχει πρόθεσμα εάν ε, η φορολογία μεταφερθεί από τις δραστηριότητε σε άλλες δραστηριότητε θα μπορέσει να συμβάλλει στις ε, πολύ αναγκαίες προσπάθειες ανάπτυξης. Επίσης βελτιώνει το οικονομικό κρυλήμα για τις επιχειρήσεις και ήθελα να τονίσω εδώ ότι είμαστε υπέρ ενός συστήματος ευρωπαϊκού για το ΦΠΑ με ξεκάθαρους κανόνες που θα δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις σε πιο προσβατή και καλύτερη ενημέρωση και δημιουργώντας ένα νέο βήμα ΦΠΑ όπως το λέμε και στη σχετική μας ανακοίνωση για ένα νέο καθεστώς ΦΠΑ. Υποστηρίζω την πρόταση όσον αφορά την ε, κοινή παγιωμένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων γιατί αυτό θα μπορέσει να μειώσει το διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία για τις εταιρείες, ιδίως μικρές εταιρείες που δρούν διασυνοριακά. Έτσι θα αποφευχθεί η διπλή φορολογία και οι διακρίσεις. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να συγχαρώ στη CB. Η Κομισιόν προτίθεται να εξτάσει καλύτερα το δομικό για δεσμευτικούς ε, μηχανισμούς όσον αφορά το θέμα τη διπλή φορολογία. Τον έφερα πολύ από εσά. Η Κομισιόν δεν έχει όμω σαν στόχο να διευκολύνει τη ζωή των επιχειρήσεων και να του δώσει κάποια πλεονεκτήματα. Στο σημερινό οικονομικό κλίμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα τη ε, τριβής ε, της ε, φορολογικής βάσης των κρατών μελών. Και έτσι εδώ έχουμε τις ε, προσπάθειες ε, καταβάλει για την καταμολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης, αλλά και της αποφυγής της διπλής φορολογίας. Η Κομισιόν σύντομα θα εξετάσει το θέμα της διπλής φορολογίας ε, σε ένα σεμινάριο για να μπορέσει να δει ποιε θα είναι οι λύσεις οι οποίες θα πρέπει να καταλήξει. Επίσης η Κομισιόν ε, να λαμβάνει περιττέρω πρωτοβουλίες για να εξτάσει το θέμα των φορολογικών παραδείσεων, της διπλής φορολογίας ε, κλπ. Επίσης ε, χαιρετίζω την ε, υποδοχή που δώσατε στην προσπάθειά μας για να αποφύγουμε τη διπλή φορολογία για τους διαμεθοριακά εργαζόμενους. Αξιότιμοι βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, όπω βλέπετε, η στάση τη Κομισιόν αντικατοπτρίζεται σε αυτέ τι γραμμέ, ευθυγραμμισμένη με την έκθεση του εισηγητή, καθώ επίση και τι παρατηρήσει που ακούστηκαν. Και χαίρομαι που βλέπω ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την ανάγκη για μια νέα ε, ευθυγραμμισμένη και συντονισμένη φορολογική πολιτική για να ξεφύγουμε από την κρίση και να προσφέρουμε στους πολίτες ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank, Frau Kommissarin Georgieva. Die Die Aussprache ist damit geschlossen. Abstimmung... Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Ε, η εξέταση θα γίνει στο 12, η ψηφορία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η επόμενη σημεία είναι ο Δημοσιονομικός Λόγος Ανθρωπιστικής Βοήθειας του, του κυρίου Έρν Χάουζα. Θα ήθελα να του δώσω το λόγο.